Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να αρχίσουμε γιατί στις 9.30 θα έρθει ο Επίτροπος και στις 10.30 πρέπει να φύγει. Συνεπώς, ας προχωρήσουμε. Πρώτα απ' όλα ανακοινώσεις του Πρόεδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές. Δύο καλά νέα. Τέλος πάντων. Ένα, αν μη τι άλλο. Καλό νέο. Η Ιδαν Κριστίν, ε, γραμματεία από τους φιλελεύθερους, περιμένει παιδί. Να, για τα τέλη Αυγούστου. Να, ένα καλό νέο. Η κυρία Σαρακιάνη είναι πρόεδρος ε, του Συμβουλίου κάπου στην Τριέστη. Η περιφέρεια έχει ένα πολύ μακρύ όνομα και δεν μπορώ να το προφέρω. Εν πάση περιπτώσει θα είναι πρόεδρος εκεί γύρω στην Τριέστη. Αυτά. Τώρα, για τους συντονιστές, τι έγινε χτες. Ορισμός εισηγητών. Έχουμε την πρόταση για οδηγία σχετικά με τις ανώτατες διαστάσεις οχημάτων που κυκλοφορούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα επιτρεπόμενα βάρη. Οι σοσιαλιστές το αναλαμβάνουν. Έπειτα πρόταση για την ετήσια χρηματοδότηση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στη θάλασσα και την ρήπανση από τα πλοία. Η πράσινη. Μη νομοθετικές εκθέσεις τώρα για την προστασία των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης. Είπαμε ότι δεν θα αναλάβουμε δράση. Επίσης όσον αφορά την εφαρμογή των στόχων 6 της ε, Πολιτικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ασφάλεια την Οδική, οι συντονιστές συστήνουν να ετοιμάσει ο Πρόεδρος προφορική ερώτηση με ψήφισμα. Γνωμοδοτήσεις. Υπάρχουν διάφορες γνωμοδοτήσεις για αποφάσεις. Γρήγορα θα σας τα πω. Ε, επιθεώρηση διαστήματος και ε, χώρου μάλλον και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επίσης στρατηγική για τη διαχείριση πλαστικών στο περιβάλλον, αθέμητες εμπορικές πρακτικές προστασία των καταναλωτών εσωτερική αγορά, κοινέ προδιαγραφές για το ΕΣΥΕΦ, e συνοχή, γεωργία, Επίσης όσον αφορά τις ε, γρήγορες ηλεκτρονικές επικοινωνίες, πράσινη βίβλος για την μακροπρόθεση χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως επίσης και ε, να ξέρετε ότι η Επιτροπή Οικονομική θα κάνει έκθεση, εμείς θα κάνουμε γνωμοδότηση, έτσι. Βέβαια, αν δεν κάνουν έκθεση, τότε εμείς δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε και γνωμοδότηση. Έπειτα, πλαίσιο 2030 για το κλίμα και τις ενεργειακέ πολιτικές. Δεν θα κάνουμε τίποτα. Ε, έκθεση ελέγχου για την Κροατία και για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την περιοχή του Δούναβη. Επίσης, κατευθύνες γραμμές και οικονομικά κίνητρα για καθαρή ενέργεια, δεν κάνουμε τίποτα. Και τέλος η κυρία Μουσκαρντίνη έχει ψήφισμα βάσει του κανονισμού 120, το άρθρο μάλλον 120 του κανονισμού, για τυποποίηση δικτύων ε, για τις ε, άδειε που δίνονται για άτομα με αναπηρίες. Η Επιτροπή, έτσι κι αλλιώς, θα ασχοληθεί και κλεισμένο το θυρών στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας είχαμε και το Συμβούλιο και τελικά δεν ήταν ε, ότι καλύτερο γιατί καταλήξαμε να συζητάμε τις διαπραγματευτικές μας στρατηγικές. Οπότε οι συντονιστές είπαν ότι ό,τι feedback έχουμε όσον αφορά τους τριμερείς διαλόγους θα γίνεται μεν σε ολόκληρη την Επιτροπή μας αλλά και κλεισμένο το θυρών. 18 Ιουνίου επίσης αποφασίστηκε ακρόαση και θα καλύψουμε οργανώσεις δύο από αεροπορικές εταιρείες, δύο από συνδικάτα και δύο από την πολιτική αεροπορία από του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, η Επιτροπή θα έρθει σε μια επόμενη συνάντηση συντονιστών για να μας ενημερώσει για την κατάσταση. Για το πακέτο τώρα για τα αεροδρόμια οι συντονιστέ αποφάσισαν να ψηφίσουμε τη διαπραγματευτική εντολή, κάτι το οποίο θα κάνουμε σήμερα. Εξωτερικές μελέτες τώρα. Οι συντονιστέ αποφάσισαν το ΕΛΚ και οι πράσινοι να επιλέξουν ε, δύο προτάσεις επιπλέον από αυτό που έχει ζητήσει ε, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Πέντε μελέτες δηλαδή θα γίνουν συνολικά. Διαρθρωμένος διάλογος με την Επιτροπή οι ομάδες θα ενημερώσουν τη γραμματεία μέχρι τις 8 Μαΐου ώστε να μπορέσει ο Πρόεδρος να απαντήσει στις ερωτήσεις του Αντιπρόεδρου Λέινε. Επιτροπολογία, η, το newsletter 7 και 8, 7 και 22 Απριλίου. Υπάρχει επίσης, το συζητήσαμε, τα διάφορα, οι συντονιστές αναφέρθηκαν στους γαλλικούς σιδηροδρόμους και περιμένουμε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ρώτησε, μάλλον η οποία έθεσε ε, σε διαδικασία ε, επί παραβάση τις γαλλικές αρχές. Ο πρόεδρος Σούλτς επίσης έχει στείλει επιστολή στον Βαρόσο και περιμένουμε αντίδραση. Επίσης, κρατικές ενισχύσεις. Οι συντονιστές αποφάσισαν να αποσυρθεί από το άρθρο 50 και η γνωμοδότηση fast track υπάρχει στα αγγλικά μόνο. Εξαιτία του χρονοδιαγράμματος δεν είχαμε αρκετό χρόνο, δηλαδή εξαιτία των διακασιών στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Και συμφωνήσαμε με ό,τι έχει συζητηθεί προηγουμένως. Αυτά έχω να σας πω όσον αφορά τους συντονιστές. Ερωτήσεις. Καλώς. Κύριε Κάντσια. Κύριε Πρόεδρε. Χθε συζητήσαμε το θέμα των κρατικών ενισχύσεων και ήμασταν ξεκάθαροι για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα ήθελα να επιμείνω λιγάκι σε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά όχι μόνο τις ενισχύσεις σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά ε, και διευρύνεται και στις υποδομές αυτός ο τρόπος, αυτό το σύστημα, κατά περίπτωση αξιολόγηση οποιαδήποτε ε, δημόσια παρέμβαση στην Ευρώπη με σκοπό να δοθεί μια νέα όθηση γενικότερα στην οικονομία. Οι κρατικές ενισχύσεις, δηλαδή, έχουν γίνει ένα είδος ε, λεμιτόμου για project τα οποία αξιολογούνται ε, μονομένα. Έχουμε την τη σε στο Μιλάνο που αν τελικά θα πρέπει να αποδώσει α, αυτά στα οποία έχουν σε αυτοί, ουσιαστικά υπάρχει το φάσμα της επτόχευσης. Το ίδιο συμβαίνει και αλλού. Ενώ δηλαδή με το ένα χέρι δίνουμε, με το άλλο χέρι ουσιαστικά ε, δυσκεραίνουμε σημαντικά οποιαδήποτε κρατική ή δημόσια μάλλον παρέμβαση. Είναι ένα θέμα επίγον και θα πρέπει να το διευκρινίσουμε το συντομότερο δυνατόν. Είναι σαφή η διευκρίνηση που ζητάτε. Χθε το συζητήσαμε με Μακρόν και η θέση της Επιτροπής είναι ξεκάθαρη επί του θέματος. Ο Πρόεδρος είπε ότι θα κάνει μια τροπολογία μίας λέξης διαγραφή, delete θα ζητήσουμε. Αυτό και τίποτα άλλο. Υπάρχει και συμφωνία της Επιτροπής ΕΚΟΝ που θα ζητήσουν τη διαγραφή. Αν κάποιοι εξημών μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ θα ζητήσουν διαγραφή τώρα το Συμβούλιο, θα ζητήσει διαγραφή, δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε για τη διαγραφή, πάντως χωρίζουμε. Πάντως αυτή η πρόταση Ξέρουμε τι συνέπειε θα έχει για τι μεταφορέ και ιδίω για τι αστικέ μεταφορέ. Σίγουρα και ο Επίτροπο το γνωρίζει. Ιδίω μετά τη χθεσινή συζήτηση. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι υπάρχει το αίτημα του άρθρου 50, το αυτό το αίτημα απεσύρθη γιατί υπάρχει διασφάλιση επιτροπής έκον. Από εκεί και πέρα εγώ δεν μπορώ να πάω παραπέρα. Ο κύριος Λίκτενμπεργκ. Κύριε. Μια παρατήρηση. Εάν δοθούν τέτοιε παραχωρήσει στην Ιταλία θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι σωστή η διάθεση αυτή. Καλώς λέει πρόεδρος, εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι το στοιχείο των δημοσίων, παρα... Παρα... των δημοσίων μεταφορών. Όχι γενικά το θέμα των κρατικών ενισχύσεων, αλλά τον επαχθούν οι μεταφορές στο... στη ρύθμιση των κρατικών ενισχύσεων είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί πολύ και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Συμφωνούμε, μάλλον δέχεστε την έκθεση πραγμένων των συντονιστών. Καλώς, αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στις ψηφοφορίες. Κύριο Σασόλη και Higgins. Άλλος κανείς. Εντάξει, θα δεχτούμε. Τα έχετε. Α, εντάξει, την έχετε. Την κάρτα σας. Λοιπόν, για να ελέγξουμε λίγο. Ψηφίστε. Δοκιμαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορία. Εντάξει, όλοι. Καλώς. Αρχίζουμε. Έκθεση Higgins. Έκθεση πρωτοβουλία στρατηγική για μια υπηρεσία τηλεδιοδίων και ένα σύστημα αυτοκόλλητων σημάτων. Παράγραφο 1, τροπολογία 12 για άλλα σέντερ. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε για την 26. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά συν μία για τα υπέρ. Ψηφίσατε όλοι υπέρ στις ψηφοφοριες εγκρινεται Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 20-19. Ο κύριος Σασόνη είναι υπέρ. Α, πήγα πολύ γρήγορα στην 25, εγώ φταίω, έπρεπε να ψηφίσουμε τη συμβαστική 2 πρώτα. Συμβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην τροπολογία 25, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26, υπέρ, κατά, αποχές, για αυτήν πρέπει να ελέγξουμε. Οπότε ελέγχουμε για την τροπολογία 26. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Συν ένα, είπαμε. Στα υπέρ. Πέρα στις φοφορίες. Τώρα απορρίπτεται. Τσίμα τσίμα. Συμβαστική τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για τη συμβαστική 5. Ο κύριος Σασόλη είναι κατά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της φοφορίας. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 και 47 μαζί για την ίδια. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 48. Ψηφίστε παρακαλώ. Ο κύριος Σασόλ είναι κατά. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ υπέρ 57 κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 3 καταπίπτει. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία αριθμός 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε καλά κύριε σας όλοι. Υπέρ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 34 υπέρ, Πέντε κατά καμία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια, κύριε Higgins. Επόμενη ψηφοφορία. Το επόμενο είναι πρόταση κανονισμού για την οδηγία 96-07 στον αφορά τα αεροδρόμια και πρόκειται για τη διαπραγματευτική εντολή υπέρ ηλεκτρονικά. Αλλά ξέρω ότι όλοι είναι υπέρ, αλλά τέλος πάντων. Ωραία, ο κύριος σας όλοι είναι υπέρ, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της πληροφορία 38 υπέρ, μία ψήφος κατά, άρα εγκρίνεται η διαπραγματευτική εντολή. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Λάκφερτ και για τον κύριο Ούγκιας. Θέλετε ξεχωριστά να ψηφίσουμε. Ωραία. Για τον κύριο Λάκφριτ, για την ηχορύπανση. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Χωριστά πρέπει έτσι κι αλλιώς να τα κάνουμε. Λάιχφριτ, ναι. Λάιχφριτ από το πακέτο για τα αεροδρόμια. Είναι η έκθεση Frit. Πέρα της φοφορίες. Και αυτός έχει την διαπραγματευτική του εντολή. Εγκρίθηκε τώρα του κύριου Ούγκιας για τις χρονοθυρίδες, τα σλότς. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Κύριε Ουγγιά, και εσείς έχετε διαπραγματευτική εντολή. Τώρα είναι η έκθεση του κύριου Κόλιτσεκ. Μία ψηφοφορία έχουμε εδώ. Κύριε Λίχτεμπεργκερ, σας ακούμε. Λυπάμαι. Πρόεδρε, σήμερα κάπως υποφέρει η ακοή μου. Είχαμε μια διαφορετική σειρά υπόψη. Θεωρούσαμε ότι ψηφίζουμε τις, χρονοθυρίδες τώρα και γι' αυτό και υπερψηφίσαμε. Αυτό είχε προβλεφθεί ως πρώτο. Και επειδή πράγματι δεν ακούω καλά σήμερα, κατάλαβα λάθος, Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω για την ομάδα μας μια διόρθωση της ψηφοφορίας. Είμαστε κατά της εντολής σας άρα. Θα το σημειώσουμε. Εντάξει, το αποτέλεσμα βέβαια της ψηφοφορίας δεν τροποποιείται με αυτό. Και η κυρία Λίχτεμπέργκερ, θα μπορούσαμε να είχαμε ψηφίσει μαζί όλες τις διαπραγματευτικές εντολές. Τις κάναμε χωριστά, με πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει εγκρίθηκε με ενισχυμένη πλειοψηφία μάλιστα η διαπραγματευτική εντολή. Τώρα έκθεση Κόλιτσεκ. Πρόκειται για απόφαση σχεδίου του Συμβουλίου για εντατική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της αεροναυτιλίας. Πρόκειται για ένα γενικό πλαίσιο συνεργασίας, ενισχυμένη συνεργασία. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Ωραία. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες και περιμένουμε τον Αντιπρόεδρο Κάλλας τώρα. Να επαναλάβω ότι έχουμε τον Αντιπρόεδρο εδώ μέχρι τις 10 και μισή. Καλό θα ήταν λοιπόν να προσπαθήσουμε να είμαστε συνεκτικοί και συμπυκνωμένα να λέμε ότι έχουμε να πούμε. He's blocked in traffic, so... Five minutes, thanks. Θα καθυστερήσει πέντε λεφτά γιατί λόγω του κυκλοφοριακού έχει μποτιλιαρίσματα. Okay, colleagues, bring you back to order, please. Και συνάδελφοι, παρακαλώ, πάρουμε τις θέσεις μας. Το επόμενο σημείο της ημερήσης διάταξης για μία ώρα, επαναλαμβάνω, είναι η παρουσίαση που μας κάνει ότι πρόεδρος Κάλλας και την οδηγία περιβαρών και διαστάσεων των οχημάτων. Λοιπόν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, θέλω να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπή Κάλλας και να του δώσω το λόγο. Καλημέρα σα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη. Πριν από μία εβδομάδα η Επιτροπή έθεσε μια πρόταση που επιτρέπει τους κατασκευαστές φωτιγών να δημιουργήσουν το φωτιγό του μέλλοντος. Αυτό αποκρίνεται στις πιεστικές κοινωνικέ προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, την οικονομική αποτελεσματικότητα και την οδική ασφάλεια. Εκατομμύρια φορτηγών θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τους δρόμους μας κάθε μέρα. Είναι προς το συμφέρον όλων μας, αναμφίβολα, καθένα από αυτά τα φορτηγά να χρησιμοποιεί λιγότερα καύσιμα, να ρηπαίνει λιγότερο και να είναι όσο γίνεται πιο ασφαλές. Ένα τούβλο είναι μάλλον το ελάχιστο δυναμικό το λιγότερο μοναδρονομικό αντικείμενο που μπορείτε να φανταστείτε. Γι' αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το σχήμα των φορτηγών του κλειστού δρόμου μα. Τα φορτηγά θα μπορούν πλέον να έχουν μια στρογγυλωμένη καπίνα μπροστά και ένα δυναμικά πτερήγια ε, πίσω. Αυτό θα καταστήσει τι οδικέ μεταφορέ πιο καθαρέ. Θα εξοικονομήσει πάνω από 7,8 τόνου ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ετησίω για μια τυπική διαδρομή φορτηγού μακρές ε, απόσταση που καλύπτει 100.000 χιλιόμετρα και ταυτόχρονα αυτό θα μειώσει ε, τις τιμές που πληρώνουν σε καύσιμα οι πράκτορες χερσαίων μεταφορών και αυτό τι σημαίνει ότι το ίδιο φορτηγό μακρά απόσταση που καλύπτει 100.000 χιλιόμετρα θα εξοικονομεί 5.000 ευρώ το χρόνο σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Και εγώ ω ποδηλάτη, μπορώ να σα πω ότι το να στέκομαι δίπλα σε ένα φορτηγό σε ένα σταυροδρόμι μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο. Όταν στρίβει ο οδηγό του φορτηγού δεξιά ή αριστερά στον βασίλειο μπορεί να μην δει τον ποδηλάτη. Γι' αυτό το λόγο η καλύτερη ε, προ προς τα πλάγια είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός νέου κανόνες για την ασφάλεια και για τα πράσινα φορτηγά που στέλνουμε. Επίσης, πέρα από την καλύτερη ορτότητα, οι νέε καμπίνες οδηγού θα έχουν μία και καμένο μάλλον σχήμα, ένα σχήμα το οποίο θα επιτρέπει να αποτρέπουμε τέτοιου είδους ατυχήματα σε πεζούς και ε, πεδιλάτες. Και επίσης, με αυτόν τον τρόπο, ε, μπορούμε να μειώνουμε κατά με τοπικών συγκρούσεων. Συνολικά αυτή η πρόταση μπορεί να μας βοηθήσει συνολικά να σώσουμε τι ζωε 300 300-500 πεζών και ποδηλατών κάθε χρόνο. Κυρίε και κύριοι, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστέ φορτηγών είναι ηγέτε στην παγκόσμια αγορά. Ο ίδιο ο κλάδο είναι βασικό επενδυτή στο τομέα τη έρευνα και τη ανάπτυξη και συνολικά οι εταιρείε φορτηγών απασχολούν πάνω από 6 εκατομμύρια εργαζομένων. Η πρόταση αυτή θα δώσει στου Ευρωπαίου κατασκευαστέ ε, μια νέα όθεση για να ξεκινήσουν να σχεδιάζουν πιο πράσινα και ασφαλή φορτηγά για να ανταποκριθούν στι απαιτήσει αγορά στο μέλλον. Είναι μια βιομηχανική ευκαιρία που θα στηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασία στην Ευρώπη και την οικονομική ανάπτυξη. Τέλο, έχω καλά νέα και για την κατάσταση των δρόμων μα. Σε κάποια κρατημέλη έω το 1 τρίτο των οχημάτων ταξιδεύουν υπέρβαρα. Αυτό οδηγεί, δημιουργεί βλάβες και ζημίες στις υποδομές, ε, δημιουργεί πρόβλημα στην οδική ασφάλεια και στρέφει στον ανταγωνισμού ανάμεσα σε εκείνους που ακολουθούν τους κανόνες και εκείνους που δεν τους τηρούν. Οι προτάσεις συμπεριλαμβάνουν συστήματα στάθμισης υψηλής τεχνολογίας που θα επιτρέπει να εφαρμόζονται κανόνες πιο αποτελεσματικά και ε, συνεκτικά σε όλη την Ένωση. Και έτσι λιγότερα υπέρβαρα φορτηγά σημαίνει και λιγότερες λακκούβες για εμάς τους υπόλοιπους οδηγούς. Έπειτα, η δυσμυρική χρήση ε, μικρών φορτηγών. Θέλω να επισημάνω ότι αυτή η πρόταση έχει στόχο τη βελτίωση της ε, απόδοσης σε θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας ε, και βιομηχανικής αν θέλετε, απόδοσης ε, των φορτηγών. Και αυτή η πρόταση δεν αλλάζει τις βασικές αρχές του κεκτημένου που επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν μεγαλύτερα φορτηγά να κυκλοφορούν στην εθνική επικράτεια των κρατών μελών. Αυτό είναι επιλογή του κάθε κράτους μέλους και παραμένει επιλογή του κάθε κράτους μέλους. Πριν από δύο χρόνια η Επιτροπή έλαβε ένα αίτημα να διευκρινίσει τι γίνεται. Αν δύο κράτη-μέλη επιτρέψουν να κυκλοφορούν αυτά τα φορτηγά στην επικρατεία τους, μετά μπορούν να περάσουν τα σύνορα. Οι νομικοί εμπειρογνώμονες Πελέθαν το θέμα και τελικά γνωμοδότησαν ότι σε αυτή την περίπτωση μπορούν να, να κάνουν τη διέλευση των σύνορων ανάμεσα στα δύο αυτά κράτη-μέλη και η Κομισιόν προέβη στην εξή διευκρίνηση σε μία επιστολή ε, που συνέταξε πέρυσι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εσείς κυρίες και κύριοι, Είστε της γνώμης ότι η διευκρίνηση αυτή μόνο με μία επιστολή δεν είναι αρκετό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει λόγο εν προκειμένου. Και αυτή λοιπόν η διάταξη θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε μία νομική πρόταση. Αυτό λοιπόν κάνουμε τώρα και βλέπετε να συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την ομιγή μας πρόταση αυτή η διάταξη. Οπότε κυρίες και κύριοι, εν κατακλείδη. Πρόκειται μια πρόταση προ όφελο όλων. Χαμηλότερε εκπομπέ ρήπων και περισσότερη ασφάλεια για την κοινωνία. Χαμηλότερα λειτουργικά ε, λειτουργικές διαπάνες ε, για τους πράκτορες αρχιστών μεταφορών και χρήστες των υπηρεσιών μεταφοράς και μια βιομηχανική ευκαιρία για όλους τους Ευρωπαίους κατασκευαστές σχήματων. Ευχαριστώ ε, τον Επιτροπό, λοιπόν, οι συντονιστές Γκρός, Αλκατράου, Μάιστερ, Λίκτενμπέρκερ, και Φώστερ. Είναι οι συντονιστές. Έπειτα, οι υπόλοιποι ομιλητές. Mr. Mrs. Mr. Ertug, Mr. Mr. Ferber, Mr. Anybody else Άλλος κανείς που θα ήθελε να μπει στον κατάλογο των αγορητών. Αυτό Okay. Αυτός λοιπόν ο κατάλογος αγορητών, λοιπόν, προτείνω να δούμε υπόψη και το χρόνο για να μπορέσει να απαντήσει και ο Επίτροπος. Τέσσερα λεπτά στους συντονιστές και τρία λεπτά στους υπόλοιπους ε, ομιλητές. Κύριε Γκρός, τέσσερα λεπτά. Και θα βάλω και το ρολόι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η πρόταση σημερινή θα οδηγήσει σε αρκετά ενδιαφέρουσες συζητήσεις, πιστεύω. Και φαντάζομαι ότι θα παρατηρήσετε και στο μέλλον, θα ακούσετε και στο μέλλον ότι και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ως πολιτική ομάδα έχει στο εσωτερικό του διαφορές. Βεβαίω θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα των πολύ μεγάλων φορτηγών, των Giga Liner όπως ονομάζονται, και ε, λύσεις εναλλακτικέ. Πιστεύω λοιπόν ότι η νομοθεσία του 96 ήταν καλό να ε, αναθεωρηθεί, να επικαιροποιηθεί, δεδομένου ότι υπάρχουν και νέες εξελίξεις, ε, δυνατότητα για την εξοικονόμηση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, η δυνατότητα για βελτίωση της ασφάλειας. Όλα αυτά είναι θετικά και πιστεύω ότι θα πρέπει να χαθούν μέσα στον όλο δημόσιο διάλογο τα δύο αυτά σημαντικά θέματα. Σε αυτά θα πρέπει να επικεντρωθούμε και όχι σε άλλα. Επίσης, απαραίτητο είναι να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου σε ένα θέμα στο οποίο η ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή με τι άλλο μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση. Είναι καλό να καταγράφονται σαφώς οι θέσεις και τώρα το Κοινοβούλιο και βέβαια μετά τα κράτη-μέλη θα, θα κληθούν να πούν εάν δέχονται να κυκλοφορούν τα mega liners στους δρόμους τους με την έγκριση ή όχι αυτού του κανονισμού. Ε, επίσης, τα διάφορα κράτη της Ευρώπης έχουν και πολύ διαφορετικές εμπειρίες. Σημειώσει, ε, έχουμε πολύ θετικές εμπειρίες στα βόρεια κράτη, στα κράτη της Βόρειας Ευρώπης και ίσως δεν υπάρχει λόγος να, ή εν πάση εγώ δεν βλέπω λόγο να απαγορευτεί κάτι το οποίο λειτουργεί ικανοποιητικά σε κάποια κράτη επειδή κάποια άλλα κράτη δεν θέλουν και δεν θέλουν να εκτεθούν στον ανταγωνισμό θα πρέπει να βοηθήσουμε, εγώ πιστεύω, σε έναν καλό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών και μπορώ να σα δώσω παραδείγματα από, επιμέ... από συγκεκριμένε εταιρείε, επιχειρήσει, οι οποίε αρχικά είχαν ταχθεί κατά τη λύση, ε, όταν όμω μπόρεσαν να εισαγάγουν στι δομέ του τέτοιου είδου φορτηγά τότε άλλαξαν στάση και άρα ίσως αυτό αποτελεί μια ένδειξη για το πώς θα ε, εξελιχθούν οι αντιπαραθέσεις μας. Βασική γραμμή πάντως πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι η ασφάλεια και υποδομές. Βάσει αυτών θα πρέπει να δίδεται η αδίποτε άδεια. Και δεν πρέπει από την άλλη η Ευρώπη να καταστεί υπεύθυνη για κάτι στο οποίο σε τελική ανάλυση θα δώσουν το πράσινο φως στα κράτη-μέλη. Είναι κάτι το οποίο και από την ανακοίνωση μπορεί να προκύψει σαν εντύπωση ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προάγει κάτι το οποίο όμως τα κράτη-μέλη μπορεί να παρεμποδίσουν ή δεν θέλουν κτλ. Αυτό λοιπόν ξεκάθαρα πρέπει να ε, δηλωθεί. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ασφαλώς θα πρέπει να κάνουμε την προσπάθειά μας για την εξέβριση μιας ενιαίας γραμμής μέσα στην πολιτική μας ομάδα. Η επικουρικότητα ασφαλώς, όπως αναφέρατε και εσείς, θα μας διευκολύνει το έργο. Ευχαριστώ κύριο Σαλκαντράουι, Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αρχίζοντας, θέλω να πω ότι από το 96 έχουμε την νομοθεσία όσον αφορά το βάρος και τις διαστάσεις των οχημάτων. Έχουν υπάρξει εξελίξεις, έχουν γίνει έρευνες, έχει τροποποιηθεί τεχνολογία. Σίγουρα υπάρχουν πολλά θετικά στην πρόταση. Το θέμα της ελαστικότητας, ευελιξίας, η δυνατότητα να ανασχεδιαστεί η καμπίνα του οδηγού, να υπάρξει ένα σχεδιασμός πιο αεροδυναμικών φορτηγών τώρα. Το θέμα της μείωσης του όγκου των καυσίμων, όλα αυτά είναι θετικά. Το ότι επίσης λαμβάνεται υπόψη το ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ηλεκτρικά ε, φορτηγά Όλα αυτά είναι θετικές εξελίξεις. Όπως επίσης και το θέμα του βάρους είναι πολύ σημαντικό για τη συντήρηση των ε, δρόμων μας, του οδοστρώματος. Και βέβαια το θέμα του ανταγωνισμού. Όλα αυτά, σίγουρα η ομάδα μου τα βλέπει πολύ επικοδομητικά και με αυτό το βλέμμα θα τα εξετάσει. Τώρα υπάρχουν όμως και κάποια άλλα. Το θέμα του εκοκόμπι, τα gigaliners. Δεν είμαστε υπέρ στην ομάδα μου για την χρήση τέτοιων ε, φορτηγών και δεν πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τον ανταγωνισμό γιατί τελικά έτσι θα έχουμε νέες προδιαγραφές στην Ευρώπη που εδώ ακριβώς στην Ευρώπη θα είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουν γιατί θα πρέπει να προσαρμοστεί η υποδομή και θα οδηγήσει σε περισσότερη ανασφάλεια στους δρόμους. Γι' αυτό και δεν θέλουμε να δοθούν κίνητρα για τέτοια φορτηγά. Σε εθνικό επίπεδο Βέβαια εννοείται ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει κάθε χώρα, αλλά δεν θα θέλαμε να διευρυνθεί αυτό. Θα θέλαμε να περιοριστεί. Θα μπορούσε να γίνει μια συμφωνία διασυνοριακά μεταξύ δύο χωρών, δεν λέω, αλλά υποθέστε ότι μεταξύ της χώρας Α και Β υπάρχει μια τέτοια συμφωνία και μετά ανάμεσα στη χώρα Β και τη χώρα Γ και μετά τη χώρα Γ και τη χώρα Δ. Τελικά θα υπάρχει μια ολόκληρη διαδρομή στην Ευρώπη όπου θα μπορούν να κυκλοφορούν τέτοια κοκόμπι ή γιγαλάινερς. Με την πρόταση αυτή είναι αυτό εφικτό ή εσείς θα πείτε όχι μόνο μεταξύ δύο χωρών και όχι μεταξύ περισσότερων. Τέλος, η νομοθεσία για τα διόδια. Προς το παρόν, το εξωτερικό κόστος και το κόστος της υποδομής είναι μεγαλύτερο εξαιτία τέτοιων φορτηγών. Πώς θα υπολογιστεί. Εσείς τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μάσινερ εκ μέρους των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτρεπε για την παρουσίαση αυτής της πρώτης νομοθεσίας. Σε πρώτη φάση βεβαίω συμφωνούμε. Είναι καλό εάν μπορεί να αλλάξει η καμπίνα οδήγησης, εάν μπορεί να είναι πιο αεροδυναμική η τομή της και ο κυρίως εάν ε, μπορούμε να έχουμε πιο ασφαλείς, λιγότερο επικίνδυνες για τον ε, ποδηλάτη ή τον πεζό καμπίνες στα φορτηγά. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ε, βέβαια θα γίνει ίσως λίγο πιο μακρύ προς τα μπρος το φορτηγό με αυτή τη μετατροπή, αλλά θα είναι πάντως ασφαλέστερο. Άλλο ένα θέμα σημαντικό είναι αυτό των εκπομπών, ανάλογα με το αν χρησιμοποιεί βενζίνη ή πετρέλαιο το φορτηγό, είναι σημαντικό να εξοικονομούμε από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ε, από την άλλη λέγεται ότι θα πρέπει να γίνει πιο μακριά η πλατφόρμα του φορτηγού έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις διεθνείς προδιαγραφές των εμπορευματοκιβωτίων που είναι ακριβώς 15 εκατοστά μακρύτερα και άρα δεν μπορούν να τοποθετηθούν σωστά πάνω στην πλατφόρμα. Ας είναι, εάν πρόκειται να προσαρμοστούμε στις διεθνείς προδιαγραφές Για τα μεγάλα φορτηγά υπάρχουν πολύ διαφορετικές ε, θέσεις. Έχουμε δει εμείς στην κάτω σεξονία από την οποία προέρχομαι με πρώτες δοκιμές ότι όπου δόθηκε η σχετική άδεια και αυτό βέβαια το οφείλουμε στους Σκανδιναβούς οι οποίοι άλλαξαν νοοτροπίες με την εισαγωγή πρώτη των μεγάλων αυτών φορτηγών όταν δηλαδή έγινε αποδεκτό ότι μπορεί ένα κράτος μόνο, μόνο του για το ιστορικό του να δεχθεί μια τέτοια λύση. Είδαμε λοιπόν ότι ε, αντί για δύο φορτηγά χρησιμοποιούνταν μόνο ένα με αποτέλεσμα να ευνοηθεί και η προστασία του περιβάλλοντος. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί οι σοσιαλιστές δημοκράτες και οι πράσινοι τάσσονται τόσο απερίφραστα κατά αυτών των λύσεων. Εδώ δεν υπάρχει κίνδυνος ε, να χαθεί η προτίμηση προς τη σταθερή τροχιά της ε, κυκλοφορίας, της μεταφοράς των ε, εμπορευμάτων. Αυτή η προτίμηση διατηρείται. Δεν υπάρχει λόγος να το φοβούνται αυτό οι φίλοι σοσιαλιστές ή πράσινοι. Παραμένει αυτή η προτίμηση λοιπόν. Από την άλλη, αν κατάλαβα καλά, εάν υπάρχει μια διοδότηση μεταξύ δύο κρατών, ε, θα μπορούν μεταξύ αυτών των δύο, από την, δηλαδή διαβαίνοντας ένα σύνορο, να κυκλοφορούν. Γιατί όχι δύο σύνορα όμως, εφόσον υπάρχουν ε, αντίστοιχα σχέσεις μεταξύ τριών κρατών διαδοχικών, όπως και ο κύριος Αλκατράοε. Ίσως είναι καλό και αποτελεσματικό εν τέλει να προχωρήσουμε και να βελτιώσουμε τις μεταφορές στην Ευρώπη. Όχι σε όλα βέβαια τα ε, τμήματα του οδικού δικτύου σε συγκεκριμένα μόνο τμήματα με συγκεκριμένες διαδρομές. Πρέπει να επισημάνουμε δε ότι είναι πιο ασφαλή από άλλα, από άλλα φορτηγά αυτά τα Giga γιατί έχουν ειδικά συστήματα ε, πέδησης, άρα ε, σταματούν πολύ πιο γρήγορα και χωρίς δυσκολία από ό,τι τα παραδοσιακά φορτηγά. Ένα άλλο πρόβλημα θα είναι ασφαλώς η εξέβρεση θέσεων στάθμευσης για αυτά, γιατί θα χρειάζονται πολύ μεγαλύτερο χώρο. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν τα 25 μέτρα με 84 ενδεχομένω τόνου, όπω αναφέρεται, μπορεί να έχουν κάποια επίδραση στι υποδομέ. Γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μα απασχολεί ιδιαίτερα, το πόσο μπορεί να επιβαρυνόνται οι υποδομέ οι οδικέ. Η κυρία Λίχτενμπεργκερ. Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κάποια στοιχεία τη προτάσεω βεβαίω μπορώ να τα υποστηρίξω, αλλά βλέπουμε ότι θα πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια και να γίνει, ε, φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια και να γίνει αποδεκτό κάτι το οποίο δεν θα ήταν διαφορετικά αποδεκτό για τις αεροδυναμικές καμπίνες βεβαίως αν αυτό βοηθήσει στο να εξοικονομήσουμε καύσιμα γιατί όχι αλλά από την άλλη δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να δώσουμε ε, θα μπορούσαμε να υποχρεώσουμε έναν παραγωγό ή έναν ε, επιχειρηματία των μεταφορών να αλλάξει στόλο και να μεταφέρει τον στόλο του σε αυτή τη νέα τεχνολογία. Άρα κάποιο σύστημα κινήτρων θα πρέπει να προβλεφθεί. Και επίσης εφόσον ε, λύουμε το ζήτημα της νεκράς γωνίας που έχει ήδη θεωρητικά λυθεί εδώ και καιρό με άλλες λύσεις δεν βλέπω ποιο είναι το πρόβλημα γιατί μιλάμε για νεκρά γωνία. για τους αισθητήρε βάρους Μακάρι, αν και με απεσιόδειξη σε σχέση με τα κράτη-μέλη, έχουμε στο θέμα αυτό τριμερή διάλογο με τα κράτη-μέλη και έχουμε με πολύ μεγάλη δυσκολία ε, έχουμε αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες δυσκολίες ακόμη και για το θέμα του ταχογράφου. Δεν ρωτώμε λοιπόν πώς μπορούμε να περιμένουμε ότι θα προχωρήσει η συζήτηση. Και περνώ στο πιο κρίσιμο σύντημα το ζήτημα των, ε, της μάζας των εμπορευματοκιβωτίων που μπορεί, ή του όγκου που μπορεί να μεταφέρει ένα εμπορευματοκιβώτιο το οποίο, για το οποίο προβλέπεται ότι μπορεί να δοθεί μια εξαίρεση ανάλογα με το εάν εξυπηρετούνται οι συνδυασμένε μεταφορές. Άρα λοιπόν εδώ μας δίνεται η δυνατότητα να επαναφέρουμε τα φορτία από την σταθερή τροχιά στους δρόμους, πράγμα το οποίο βεβαίως προφανώς και μας ενοχλεί. Για τα Gigaliner και την διασυνοριακή διάβαση από πλευρά τους των ε, τη διασυνοριακή κυκλοφορία θα μιλήσει ο κύριος Κράμερ αλλά το σημαντικό είναι εδώ ότι ε, η ερμηνεία από πλευρά του Κοινοβουλίου είναι σαφής Με το greenwashing αυτό το οποίο προσπαθείτε να μας περάσετε, ταυτόχρονα προσπαθείτε να μας κάνετε να καταπιούμε το πιο δύσκολα, το, τα, τα Giga Liner δηλαδή, γιατί βλέπουμε ότι ε, θα ασκηθεί πίεση από τα κράτη τα οποία τα προτιμούν με όποιες απειλές μπορούν οι εμπάσχευτος μέσα πίεσης και στα υπόλοιπα που δεν τα θέλουν να τα δεχθούν. Ε, επαναλαμβάνω, μόνο οι επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν τα gigaliner έχουν ε, από αυτά πλέον εκτήματα και μόνο σε επίπεδο κόστους. Ούτε για τις υποδομές, ούτε για το περιβάλλον, ούτε για τίποτε άλλο προσφέρουν τα gigaliner. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι εάν γίνει καλύτερη κατανομή του βάρου στον άξονα, νομίζω ότι λύνεται το πρόβλημα της επιβάρυνσης των υποδομών, των οδικών υποδομών, χωρίς να χρειάζεται να περάσουμε στα Gigaliner. Είναι για μένα λοιπόν πολύ αμφιλεγόμενη αυτή η πρόταση. Γιατί βλέπω ότι προσπαθεί να εισαγάγει νέες διαστάσεις, γίγκα, λάινερ, μεγάλες διαστάσεις, τάχα ως πλεονέκτημα για τις οδικές μεταφορές και να μας κάνει να καταπιούμε αυτή τη λύση από το Κοινοβούλιο. Αυτό κρύβεται πίσω από την πρόταση. Ευχαριστώ. Foster is your. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ. τον κύριο Επίτροπο θέλω να πω ότι συμφωνώ με κάποια από τα σχόλια των συναδέλφων. Η αλήθεια είναι ότι λάβαμε αυτό το κείμενο τελευταίε μέρε, οπότε χρειαζόμαστε να το μετρήσουμε σε μεγαλύτερο βάθο. Πάντω, γενικώ, πώ κανεί θα διαφωνούσε σε αυτή την πρόταση. Έχουμε πιο προηγμένε τεχνολογίε, ε, πιο καθαρά περιβαλλοντικά και πιο ασφαλή φορτηγά. Αλλά ε, ρωτώ, το πρώτο μου ερώτημα είναι, έχει γίνει συζήτηση με του σχεδιαστέ. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι σχεδιαστή των φορτηγών, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε να πάρουμε μια κάποια ιδέα. Τι λέει ο κατασκευαστικό κλάδο, τι δυνατότητε ε, υπάρχουν και με τη χρονοδιάγραμμα. Γιατί μπορούμε να το συζητάμε όλη τη μέρα αυτό το θέμα, αλλά το θέμα είναι αν τελικά προχωρήσουμε για την πρόταση, πρέπει να ξέρουμε τι μπορούν να κάνουν οι κατασκευαστέ. Πρώτο ερώτημα. Ε, συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Μάισνερ σχετικά με τα μεγαλύτερα φορτηγά Δηλαδή κάποιε φορέ αυτό το επιχείρημα κάποιων δεν το καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι μικρά τα φορτηγά γιατί άμα είναι μικρότερα ε, θα είναι πιο πολλά στου δρόμου. Κάπου πρέπει να βρούμε μια συμφωνία. Να κάνουμε ε, κάποιες υποχωρήσεις. Συμφωνώ, μεγαλύτερα φορτηγά που είναι πιο προηγμένα τεχνολογικά. Αν υπάρχει τεχνολογία θα έχει και λιγότερα φορτηγά στους δρόμου. Οπότε συμφωνώ. Θα χρησιμοποιούν λιγότερα καύσιμα. Ένα φορτηγό αντί τριών στου δρόμου. Και βεβαίω θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλε οδικέ υποδομέ για να μπορούν να τα δέχονται. Βέβαια, στον Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε κάποιο πρόβλημα στο θέμα ασφάλεια, γιατί οδηγούμε ε, ανάποδα στου δρόμου. Άρα το θέμα είναι. Το πρόβλημα είναι το θέμα του σχεδιασμού ε, λαμβάνει υπόψη και αυτή την οδήγηση και πώ ακριβώ αποφύγουμε την νεκρέ γωνίε. Ξέρω ότι δεν υπάρχει πρόθεση να μα παραγνωρίσετε, αλλά είναι καλό οι σχεδιαστές να λάβουν και αυτό υπόψη. Τώρα, για τον έλεγχο αυτών των φορτηγών. Συζητούμε γενικότερα το πακέτο για την ε, εξοπιστία των οδικών ε, αρτηριών και θεωρώ ότι εκεί πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη και ήδη λαμβάνεται υπόψη. Ήδη κάνουμε δουλειά σε αυτόν τον τομέα, στο τομέα του ελέγχου. Και αν επιτρέπετε και κάποια άλλα σχόλια, Πρόεδρε. Αυτέ οι δύο χώρε, το παράδειγμα τη δύο χώρε, αν εγώ είχα ένα φορτηγό στη Βόρεια Ιρλανδία και θέλω να πάω στην Ιρλανδία, που είναι ακριβώ στο Γιονυσί. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω. Ή το φορτηγό πληρεί του κανόνε και μπορεί βάσει των συμφωνιών να κινηθεί Ή Ιδάλω, γιατί να περιορίσετε σε μια χώρα, δεν καταλαβαίνω ειλικρινά αυτό το θέμα. Ή α, είναι αξιόπιστο να κινηθεί στους δρόμους ή όχι. Παντού όμως. Και τέλο για τον προπολογισμό. Όταν διαβάσετε την πρότασή σα παραπέμπεται στον προπολογισμό των ε, διευρωπαϊκών δικτύων. Τι σημαίνει αυτό, μπορείτε να μου καλύτερα. Και τέλος για τις μεταβατικές περιόδους για τα νέα φορτηγά που τελικά θέλουμε να αποκτήσουμε σε σχέση με τα μικρότερα φορτηγά που κυκλοφορούν σήμερα, που κάνουν μικρές αποστάσεις και τα οποία δεν θα επενδύουν πλέον ε, ενδιαφερόμενο στο μέλλον. Δεν περιμένετε όμως ότι όλοι θα ανανεώσουν ε, έτσι μια νυχτή το στόλο τους, άρα θέλουμε να μα πείτε κάτι για τη μεταβατική περίοδο. Ευχαριστώ για την πρόταση και θέλαμε κάποιε λεπτομέρειε περισσότερο ε, από αυτών των θεμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα ο συναδέλφο. Ο κύριος Πάρκερ, τρία λεπτά. Πίρκερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η πρόταση, κύριε Αντιπρόεδρε, εν γέννη, με την επεξεργασία της ε, οδηγίας του 96 βεβαίω είναι ευπρόσδεκτη. Κοιτάζοντας όμως την λεπτομέρειε τη, της, ε, πάλι είναι πολλές οι θετικές πτυχέ. Πέραν των βελτιώσεων που αναφέρθηκαν ήδη της αερονοδυναμικής για λόγου οικολογικού, τα μέτρα ασφάλειας, ε, τους καθρέφτες, εξωτερικού καθρέφτες, όλα αυτά είναι θετικά. και η όπως επίσης η δυνατότητα για την ε, διαλειτουργικότητα που θα βελτιωθεί σε σχέση με τα εμπορευματοκιβώτια των 54 ποδών. Αυτά λοιπόν έχουν μεγάλη σημασία, καλύτερη χρήση, βελτίωση της ασφάλειας και βέβαια ε, συνθήκες θεμητού ανταγωνισμού. Για τα λεωφορεία επίσης πρέπει να πούμε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση, είναι πιο καλός ο εξοπλισμός τους, είναι πιο ασφαλή. Βέβαια και το μεγαλύτερο βάρος των επιβατών θα αποτελεί ένα παράγοντα που θα πρέπει να υπολογιστεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ευπρόσδεκτες οι προτάσεις σε αυτό το βαθμό. Αλλά δεν μπορώ να χαρακτηρίσω ευπρόσδεκτη την πρόταση για τα λεγόμενα gigaliner και την αδειοδότησή τους για τη διασυνοριακές μεταφορές. Βεβαίως μπορεί κάποιο κράτος μέλος, και σε αυτό δεν έχουμε αντίρρηση, να δεχθεί για το εσωτερικό του τέτοιες λύσεις. Γιατί βεβαίως για κάποια κράτη και για κάποια διαδρομές μπορεί να είναι θετικό. Αλλά αν κοιτάξουμε στη χώρα μου την Αυστρία την κατάσταση, όπου Έχουμε μια σειρά από ε, γέφυρες, από περιφερειακούς δρόμους, από τούνελ που θα χρειαστεί να αναδιαμορφωθούν μόνο και μόνο για να χωρέσουν αυτά τα λάινερ. προφανώς δεν αξίζει τον κόπο. Και επιπλέον, εάν γίνει αυτό διασυνοριακά, αναμφίβολα θα βρεθούμε κάποια στιγμή στην κατάσταση κατά την οποία τα κράτη τα οποία με την αρχή της επικουρικότητας αποφασίσουν να μην δεχθούν τα τζιγκαλάινες για τους δικούς τους θεμητούς και σωστούς λόγους θα βρεθούν σε κατάσταση που θα τους ασκηθούν πιέσεις, διότι τα κράτη που έχουν δεχθεί εισαγάγει στο σύστημά τους τα τζιγκαλάινερ από το βορρά θα θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν για τις μεταφορές τους στο νότο και θα πρέπει να περάσουν από την Αυστρία και άρα θα είναι κατάσταση αφόρητα. Και μετά βεβαίως θα πρέπει να δούμε από τη διαδρομή α στη β, από τη β στη γ, από τη γ στη δ, πώς είναι δυνατόν να είναι λογικό το να επιτρέπεται το ε, Liner, αλλά να μην επιτρέπεται στα ενδιάμεσα κομμάτια και άρα να, πώς είναι δυνατόν να θεωρείται ότι έτσι μπορεί να ε, να, να επιτρέπεται από το ένα κομμάτι στο άλλο σε διμερεί σχέσει και τελικά να μπορεί να διαπέρνει ολόκληρη την Ευρώπη. Επομένω, η κατάσταση είναι ένα σαφέ όχι από πλευρά μα. Ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε τον Επίτροπο για την παρουσίαση αυτή. Ευχαριστούμε για την αναθεώρηση αυτή που προτείνεται της οδηγίας, κάτι που περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στόχος βέβαια της αναθεώρησης αυτής είναι να βελτιωθεί η ασφάλεια στους δρόμους. Και γι' αυτό και εμείς θα στηρίξουμε όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην ε, οδική ασφάλεια, στην βελτίωση του σχεδιασμού της καμπίνας του οδηγού και όλα τα άλλα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν ε, με το νεκρό σημείο κλπ. Τώρα, όσον αφορά το βάρος και τον ταχογράφο, εμείς θέλουμε να εισαχθούν οι αισθητήρε αυτοί για το βάρος, όμως δυστυχώ οι περισσότερε χώρε αντιτίθενται. Δεν αντιτίθενται ουσιαστικά στην ίδια την ιδέα των αισθητήρων αυτών βάρους, αλλά λένε ότι ο κανονισμός για το ταχογράφο δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να συμπεριλάβουμε την ιδέα αυτή των αισθητήρων βάρους. Εμείς, εγώ όμως θα ήθελα να υπάρξει γιατί πιστεύω ότι θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια και πιστεύω ότι θα βρούμε και την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Όσον αφορά τώρα τα μεγάλα φορτηγά, τα gigaliners, το Κοινοβούλιο το έχει συζητήσει, έχει εκφραστεί σχετικά. Για μας το πιο σημαντικό είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και πιστεύω ότι μετά την συζήτηση στο Κοινοβούλιο θα καταλήξουμε σε μία οδηγία η οποία να είναι ορθή, νομικά ορθή δηλαδή, ώστε να τελειώσει πια όλη αυτή η συζήτηση για τα gigaliners ναι ή όχι νομικά, να ξέρουμε τι ισχύει. Και είμαι πεπισμένη ότι τελικά το κείμενο θα μπορέσει σύντομα σχετικά να υιοθετηθεί και θα συνεισφέρει και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σερτού για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Είναι πολλά τα σημεία, τα στοιχεία της προτάσεως τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασία και της ασφάλειας στους δρόμους της Ευρώπης. Ξέρετε ότι αυτό είναι ένα αίτημα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί τη ζητήσει την αναθεώρηση, με την αναθεώρηση οδηγία να Ε, βελτιωθούν οι συνθήκες της ασφάλειας ε, και της ε, περιβαλλοντικής προστασίας. Ωστόσο, εσείς κάνετε μια πρόταση, κύριε Πρόεδρε, για τη διασυνοριακή κυκλοφορία των Giga Liner, τα όμως πρέπει την οποία όμως πρέπει να κοιτάξουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Εσείς λέτε στην πρόταση ότι μόνο υπό ορισμένε συνθήκες και με συγκεκριμένη προηγούμενη αίτηση μπορεί να γίνει αυτή η κυκλοφορία. Μπορείτε να μου πείτε παρακαλώ ποιο θα ελέγχει αυτές τις προϋποθέσεις, ότι τηρούνται και σε περίπτωση που παραβιαστούν οι προϋποθέσεις τι είδους κυρώσεις προβλέπετε. Γιατί δυστυχώς δεν γράφετε τίποτα για το θέμα αυτό στην πρόταση οδηγίας. Και από την απάντηση που μας είχατε δώσει στις 15 Ιανουαρίου αναφέρω ότι είχατε πει και παραθέτω ότι δίνανται τα κράτη-μέλη να χορηγήσουν τη σχετική άδεια. Αυτό το δίνανται, ξέρουμε τι γίνεται εν τέλει, σε τι μεταφράζεται. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν επαρκείς ε, έλεγχοι, όταν δεν υπάρχει επαρκείς επιτήρηση του συστήματος, προφανώς κύριε Επίτροπε υπάρχει αδυναμία να προβλέψει κανείς τις συνέπειες τη αγωγή του μέτρου αυτού, αυτό που αναφέρεται δηλαδή στο άρθρο 4. Και γι' αυτό, δεδομένου ότι είναι θετικές οι προτάσεις για το περιβάλλον και την βελτίωση της ασφάλειας στο υπόλοιπο κομμάτι των προτάσεών σας, δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω πόσο δυσάρεστο είναι το ότι δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση επιπτώσεων στο υπόλοιπο κομμάτι, στο κομμάτι που αφορά τα gig liners. Ρωτώ λοιπόν γιατί και πώς είναι δυνατόν να παραμελήσατε την πλήρη αξιολόγηση επιπτώσεων σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Διότι με τον τρόπο αυτόν Ε, μια πρόταση η οποία στα άλλα στοιχεία είναι καλή καθίσταται απαράδεκτη για τις διασυνοριακέ αυτές μεταφορές με τα Giga Liner. Γιατί λοιπόν στον τομέα των κυρώσεων, των ελεκτικών μηχανισμών δεν έχετε κάνει ε, αξιολόγηση επιπτώσεων. Ευχαριστώ κύριο Σκόχ. Ευχαριστώ πολύ Επίτροπε Κάλλας για τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας. Μια-δυο παρατηρήσεις για τα μεγάλα ε, φορτηγά θα ήθελα να πω ότι δεν είναι τέρατα, δεν είναι τα τερατώδη φορτηγά, είναι λαϊκιστικό τώρα να λέμε ότι είναι τέρατα φορτηγά. Μπορούν τα μεγάλα αυτά φορτηγά, τα μακρά φορτηγά να αποτελέσουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα για το συνολικό στόλο ενός ε, μιας μεταφορικής εταιρείας, δεν θα τον αντικαταστήσουν πλήρους. Ε, μπορεί να είναι πιο βαρεά, βαριά, αλλά μεταφέρουν περισσότερο φορτίο Πράγμα το οποίο έχει και θετικέ επιπτώσει προ την αποτελεσματικότητα αλλά και την προστασία του περιβάλλοντο. Δεύτερον, δεν, ε, ούτε είναι καν επιθυμητό, αλλά ούτε και δίνεται η άδεια να κυκλοφορήσουν τα μεγάλα αυτά φορτηγά ε, ε, σε όλε τι οδού, σε ολόκληρο το δικό δίκτυο, μόνο σε συγκεκριμένε διαδρομέ. Αλλά θα πρέπει σε αυτέ τι διαδρομέ να του επιτρέπεται η κυκλοφορία. Επίση, τα μεγάλα αυτά φορτηγά έχουν ιδιαίτερα ε, προωθημένης τεχνολογίας συστήματα ε, πέδησης, ε, οδήγησης και επομένως είναι πολύ πιο ασφαλή. Επιπλέον δε θα επικαλεστώ την αρχή της επικουρικότητας. Εάν ένα ζευγάρι κρατών μεταξύ τους επιτρέπουν την κυκλοφορία αυτών φορτηγών, γιατί θα πρέπει να αποκλειστεί γιατί θα πρέπει να είναι απομονωμένα από την ε, μεταφορά αυτή. Νομίζω ότι είναι ε, πολύ δυσάρεστο το να προσπαθεί κανείς να, να αποτρέψει ή να αποκλείσει τα κράτη από την ελεύθερη επαλλαγή. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Βέρμπερ. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πρέπει στην Επιτροπή μας, τουλάχιστον κάποιοι συνάδελφοι, να αποφεύγουμε να πέφτουμε θύματα της ε, επιχειρηματολογίας την οποία προβάλλουμε. Θα υπενθυμίσω κύριε Επίτροπε όταν ήσασταν εδώ πριν από ένα χρόνο ότι σας είχαν κατηγορήσει για το ότι θέλατε να επιτρέψετε στους Φινλανδούς και τους Σουηδούς να χρησιμοποιούν αυτά τα μεγάλα φορτηγά στις ε, μεταξύ τους ε, μεταφορές, πράγμα που έπραταν ήδη, αλλά απλώς δεν καλύπτονταν από μια ε, ευρωπαϊκή οδηγία. Εν τω μεταξύ θέλησατε και θεσπίστηκε η νομική βάση την οποία είχατε επιδιώξει εσείς, αλλά τώρα κατηγορείτε κατηγορήσετε για τη θέσπιση μια νομική βάση την οποία ζητούσαν εκείνοι που σα κατηγορούσαν τότε. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Κράμερ, για εσά είναι απλό ο κόσμο. Αλλά θα σα πω ότι είναι πολύ πιο περίπλοκο ο κόσμο από ό,τι θέλετε να τον δείτε εσεί και να τον παρουσιάσετε. Δεύτερον, ε, πρέπει να συζητήσουμε μέτρα και σταθμά και μόνο μέτρα και σταθμά. Αυτή τη στιγμή μιλούμε για όγκο και όχι για μάζα, βάρος. Ως εκ τούτου, περιοριστικός όρος είναι ο όγκος και όχι το βάρος όπως έχει αποφασιστεί. Με βάση αυτό το κριτήριο θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση και στο πλαίσιο της μάζας, στο, στο βάρος δηλαδή, μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία γιατί ε, η τεχνολογία μας έχει επιτρέψει τα τελευταία χρόνια την δυνατότητα αυτή, κάτω στο οποίο δεν παρεμβαίνει καθόλου η οδηγία. Εάν ε, εκεί στραφούμε παραδείγματι και κοιτάξουμε το θέμα της ασφάλειας της ε, φόρτωσης, δεν υπάρχουν νομοθετήματα τα οποία να ορίζουν κάτι διαφορετικό από την επιδίωξη της ε, ασφαλούς φόρτωσης για ασφαλείς μεταφορές. Βεβαίως, μπορώ στα όσα είπε ο κύριος Πίρκερ να δείξω εγώ κατανόηση στο βαθμό που δεν είναι δυνατόν τα 25, το, εάν σε κάποιο ενδεχόμενο τα 25 κράτη-μέλη από τα 27-28 αποφασίσουν να κάνουν ε, κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή να εισαγάγουν αυτά μεγάλα φορτηγά και να βρεθούν στη μέση η, ε, το κέντρο της Ευρώπης, Φερρυπίνη, Αυστριακή, Λουξεμβούργη και ίσως και οι Γερμανοί ε, και να ασκηθεί πίεση σε αυτούς για να δεχθούν αυτά τα φορτηγά. Όχι, θα είναι διμερείς οι συμφωνίες, η περιφέρεια μπορεί να κάνει διμερείς συμφωνίες και δεν μπορεί να ε, ασκήσει πίεση στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης ώστε να αλλάξουν στάση. και μέτρα, τα μέτρα και σταθμά είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό και είχαμε πει ότι μπορούν κάποια κράτη να προβούν ε, σε μια ε, αποδοχή νέων ε, λύσεων όπως τα μεγάλα αυτά φορτηγά αλλά δεν μπορούν να πιέζουν τα άλλα κράτη να ε, υποχρεωθούν να τα περάσουν. Ο κύριος Κράμερ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και ευχαριστώ πολύ για τα όσα υπόθηκαν τώρα. Θα ήθελα να πω ότι φαίνεται πως η μνήμη σας αρκεί μόνο για 365 μέρες, γιατί εγώ πριν από τρία χρόνια είχα πει ότι δεν επιτρέπεται αυτή η λύση της διμερούς ε, συμφωνίας για τα γιγαλάινερ. Ευτυχώς δεν μπορέσατε να το περάσετε και ο κύριος Βέρπερ ουσιαστικά σας δίνει απάντηση σε αυτά τα επιχειρήματα. Βεβαίως θέλουμε όλη τη μείωση λοιπόν των εκπομπών, αλλά γιατί 25 χρόνια δεν έχετε κάνει τίποτα και ακόμη και τώρα δεν έχετε κάνει τίποτα για να μειώσετε το όριο ταχύτητα στα 130 για να ε, βελτιώσετε τις συνθήκες καύσης του καύσιμου ε, επιπλέον για την ασφάλεια γιατί δεν έχετε κάνει τίποτα για τους εξωτερικούς καθρέφτες μέχρι τώρα και έρχεστε ξαφνικά με αυτές τις προτάσεις. Όταν έχουμε ένα gigaliner το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερο μήκος, πολύ μεγαλύτερο βάρος πώς είναι δυνατόν να μας μιλάτε για αύξηση των ε, ε, της ασφάλειας και επιπλέον από πού και που θα είναι επαρκείς για να βεβαιωθούμε ότι τηρούνται οι κανόνες, όποιοι είναι αυτοί. Άρα λοιπόν, με την πίεση του Κοινοβουλίου και του Προέδρου βεβαίω του Κοινοβουλίου έχουμε ε, ε, ζητήσει να γίνουν αυτέ ε, οι μελέτε, αλλά δεν κάνατε αξιολόγηση επιπτώσεων. Υπάρχουν Ινστιτούτα τα οποία έχουν πει ότι το, η εισαγωγή του Giga Liner θα σημάνει 12% μετατόπιση του φορτίου της σταθερής τροχιάς στις οδικές μεταφορές και πολλά άλλα δυσμενή ε, ε, αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε να πραγματοποιούνται με το που θα εισαχθούν με βάση προβλέψεις αυτές τα Giga Liner. Είναι πολύ σοβαρές οι πιέσεις, το ξέρουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα έχει μπορέσει με τις διμερείς μεταφορές να ασκήσει ε, πίεση στις, ε, στην Ελβετία επί παραδείγματι και να δεχθεί τελικά η Ελβετία από τους 28 τόνους ανώτατο που είχε τους 48 τώρα. Αυτό το ίδιο πράγμα θα φανεί και με τα Giga Liner. Θα ασκηθούν οι πιέσεις και θα υποχρεωθούν μικρότερα κράτη ή κράτη διέλευση να τα εγκριθούν, να τα εγκρίνουν. Άρα λοιπόν ε, μπορεί να υπάρχουν πλεονεκτήματα οικονομικά, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιου είδους συμφέροντα μόνο. Πρέπει να κοιτάξουμε το γενικό συμφέρον, το κοινωνικό συμφέρον, το συμφέρον του περιβάλλοντος. Είναι 5,5 Είναι 5,5 δισεκατομμύρια το κόστος τη ε, μετατροπής των οδών, ε, γεφυρών κτλ. που ανέφερε ο κύριος Σπίρκερ. Για τη Γερμανία διανοείστε τι είδου κόστος θα σήμαινε η αναμετατροπή του οδικού δικτύου για να μπορούν να περάσουν αυτά τα γίγα λάινερ και για ποιου του συμφέροντων. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά των οδικών μεταφορών. Δεν ε, απευθύνεται η πρότασή σα προ την κοινωνία, μόνο το ο μόνος στόχος που εξυπηρετείται είναι η, μεταφορά, η μετατόπιση του φορτίου από τη σταθερή τροχιά στην οδό, στο οδικό δίκτυο. Αυτό αντιλέγει, αντιβαίνει σε κάθε στόχο ορισμένο και αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Συναλόβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, λέει κυρία Σενάλοβα, για την παρουσίασή του και να σας πω ότι το θέμα της οδικής ασφάλειας είναι το πιο σημαντικό. Αυτό θέλω να στηρίξω και να στηρίξω μέτρα που βελτιώνουν την ε, σταθερότητα, γιατί μιλάμε και για τους ε, χρήστες. Μιλάμε επίσης για συγκρούσεις με ποδηλάτες που συχνά έχουμε τέτοια ατυχήματα με ποδηλάτες και φορτηγά. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε σοβαροί και αν εννοούμε πραγματικά αυτό που λέμε για την οδική ασφάλεια και την μείωση των σοβαρών ατυχημάτων στο Ευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο, αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Στηρίζω επίσης το θέμα για το βάρος, γιατί όπως λέτε, το 1 τρίτο των οχημάτων είναι πιο βαριά από όσο θα έπρεπε, κάτι το οποίο επηρεάζει την ποιότητα του οδοστρώματος και την οδική ασφάλεια. Όταν μιλάμε τώρα για τα Giga εδώ θα συμφωνήσω με εκείνους οι οποίοι έχουν μια επιφύλαξη όσον αφορά τη χρήση τους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στεπάκερ, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μια καλή πρόταση αυτή του Επιτρόπου γιατί μιλάει για τον εξυγχρονισμό, την καινοτομία, λαμβάνει υπόψη το θέμα του περιβάλλοντος και της ασφάλειας. Άκουσα διάφορα ζητήματα τα οποία με προβληματίζουν εμένα που είμαι πεπισμένος Ευρωπαίος. Διάφορα για τα Giga Liners, τα Eco και με εκπλήσει που εκείνοι οι οποίοι φωνάζουν για περισσότερη Ευρώπη, για μεγαλύτερη ολοκλήρωση, είναι αυτοί οι οποίοι αντιτίθενται σε αυτή την πρόταση. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν την καινοτομία, την αποτελεσματικότητα να την εμποδίζουν και συνειδητά να υποστηρίζουν μία μόνο μέθοδο. Εμείς, αντίθετα, έχουμε αποφασίσει για τις πολυτροπικές μεταφορές και όχι για έναν τρόπο μόνο μεταφορών, γιατί έτσι πιστεύουμε ότι είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Τώρα άκουσα λοιπόν τις συζητήσεις, τι λένε οι σοσιαλιστές, τι λένε οι πράσινοι, που τελικά είναι κατά της αποτελεσματικότητας της μεταφορές. και δεν θέλουν περισσότερα φορτηγά στους δρόμους. Εγώ όμως είμαι σαφής. Πιστεύω ότι πρέπει τα γίγα και τα Combis να μπορούν να κυκλοφορούν στις χώρες εκείνες όπου υπάρχει συνένεση από αυτών που τα θέλουν και που είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν και στην ασφάλεια και στις μεταφορές. Για όνομα του Θεού, γιατί θα εμποδίσουμε αυτές τις χώρες να επιτρέψουν σε αυτά τα φορτηγά να περνάνε μέσα από αυτές. Έπειτα για το θέμα τώρα του βάρους των ε, τόνων κλπ. Εγώ πιστεύω ότι με την πρόταση αυτή πρέπει να προχωρήσουμε και να σκεφτούμε τελικά τι βήματα μπορούμε να πάρουμε όσον αφορά και την αποτελεσματικότητα και για να επιτρέψουμε στον καταναλωτή να έχει την επιλογή, να επιλέξει τον τρόπο μεταφοράς και σίγουρα να επιλέξουμε διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, να το συνδυάσουμε μεταξύ τους και να μην βάζουμε φραγμούς στις εσωτερικές μεταφορές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Ευχαριστούμε. Κύριε Πίτροπε, εσείς έχετε και πάλι το λόγο. Βλέπετε ότι το 90% της ε, πρότασής σας είναι ευπρόσδεκτο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν βέβαια πολιτικές αποχρώσεις και διαφορές εδώ μεταξύ των μελών ανάλογα με την πολιτική ομάδα. Και βλέπετε ότι οι μεν κατηγορούν τους δε. Ε, συνηθισμένο αυτό. Οπότε μέσα σε αυτό το κλίμα θα πρέπει να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότυπα με του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολιτικό, πώ σίγουρα αυτή η πρόταση μπορεί να χωριστεί σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλο αφορά βελτίωση τη ασφάλεια, ε, βελτίωση τη περιβαλλοντική περιφορά και αυτό αφορά την κατασκευή των ε, φορτηγών οχημάτων. Και αυτή η πρόταση ουσιαστικά ξεκίνησε ε, ξεκινήσαμε την επεξεργαζόμαστε με το που μπήκαμε σε αυτή την θητεία ε, στην Επιτροπή στη συνεργασία και διαβούλευση με τι οικολογικέ με κυβερνητικέ οργανώσει και ιδίω με αυτού που ασχολούνται με θέματα οδικών μεταφορών. Σε ό,τι αφορά του κατασκευαστέ ή του σχεδιαστέ, αν θέλετε, των φορτηγών οχημάτων ε, που συμπεριλαμβάνονται ω συνομιλητέ σε αυτή την πρόταση, Άκουσα τις ερωτήσεις και τους αισθητήρε και για τους ελέγχους νομοθεσίας. Ναι, είναι πολύ ε, θεμητά ερωτήματα. Αλλά τα τελευταία χρόνια μπορούμε να πούμε ότι η διαστηριακή εφαρμογή της νομοθεσίας ε, του κώδικα κυκλοφορίας έχει βελτιωθεί σημαντικά και η αστυνομία με χαρά σημειώνει ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση από μία χώρα υιοθέτησε την διοσυνεριακή εφαρμογή του κώδικα κυκλοφορίας. Αυτό φορά την ταχύτητα, ζώνες ασφαλείας, κατανάλωση αλκοόλ και παραβίαση ε, του κόκκινου σηματοδότη. Αυτά τα τέσσερα βασικά ε, στοιχεία του ΚΟΚ, τα οποία πλέον ισχύουν διασυνοριακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα ε, που υπάρχει αυτή πλέον η ενιαία προσέγγιση και εκεί λύσαν υπόψη πλέον οι παράμετροι που αφορούν τα φορτηγά οχήματα και ο έλεγχος αυτών. Βεβαίω ο κόσμος δεν είναι ιδανικός και πάντοτε υπάρχει τα η κυρία Φώστα μου ρώτησε για την ε, κατασκευαστικό κλάδο και τη μεταβατική περίοδο. Μα ήδη κάποιοι κατασκευαστές έχουν όλα στα website τους ε, τα νέα ναι, αυτά φορτηγά. Μπορείτε να δείτε στο website της ΜΑΝ για παράδειγμα και να δείτε, χωρίς να βάζουμε καταληκτικές ημερομηνίε, αλλά δεν υπάρχει και μεταβατική περίοδος μέσα στην οποία ε, περιμένουν τα φορτηγά. Γιατί τα φορτηγά μπορούν να έρθουν και νωρίτερα. Αυτό έχουμε ζητήσει και εμεί. Κάποιοι κατασκευαστέ ήδη ήδη επεξεργάζονται νέα μοντέλα και με μεγάλη χαρά ε, είναι έτοιμοι να δεχτούν τη νέα μας πρόταση. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό για την αγορά και θα είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τους ευρωπαίους κατασκευαστές. Σύντομα λοιπόν θα δούμε αυτά τα νέα φορτηγά στους δρόμους βεβαίως. Τα φορτηγά ναι είναι δαπανηρά και χρειάζεται να περάσει μια 15 ετία ως 20 ετία για να γίνει απόσβεση της επένδυσης. Αλλά με το νέο αυτό περιβάλλον και τις νέες τεχνολογίες είναι ευπρόσδεκτη μετά μετάβαση σε αυτή τη νέα γενιά. Είναι καλό λοιπόν να έρθουν αυτά τα νέα φορτηγά των στομάτων των όσο νωρίτερα μπορούν να να αποκριθούν. Το δεύτερο σκέλος της πρότασης το ζήτημα το διασυνοριακό, η διασυνοριακή διάσταση. Είχαμε έντονε συζητήσει και στου κόλπου τη Επιτροπή κατά πόσο θα πρέπει να συμπεριληφθεί αυτή η διάταξη ή όχι. Και υπήρχαν και ισχυροί υποστηρικτέ θέσεων ε, κατά τη συμπερίληψη. Γιατί, τι θα σημαίνει αυτό, ότι όλα τα θετικά στοιχεία τη πρόταση θα εξανεμιστούν και θα εξαφανιστούν μπροστά στο φάσμα αυτής της διασυνοριακής, αν θέλετε, ρήτρας. Οπότε, σας ζητώ, εσείς είστε πολιτικοί, ε, ας παρακαλώ όμως να μην επιβραδύνετε τις διαδικασίες ε, για να υιοθετηθεί αυτή η πρόταση για αυτό το ζήτημα, γιατί δείτε όλα τα άλλα στοιχεία, τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς, της ασφάλειας, την περιβαλλοντική συμπεριφορά κτλ. που δίνει αυτή η πρόταση. Θυμάμαι χρόνια πριν στην ίδια αίθουσα η Επιτροπή έτυχε πολύ σοβαρών επικρίσεων, γιατί είχαμε την πρόθεση να τα διευκρινίσουμε όλα αυτά μόνο μια επιστολή και μας είπατε ότι δεν γίνονται αυτά με επιστολές πρέπει να υπάρχει μια νομοθετική πρόταση την οποία θα εξετάσει το Κοινοβούλιο. Να λοιπόν η πρόταση εδώ στο τραπέζι. Εσείς ε, το ζητήσατε και η Επιτροπή Μεταφορών να ζήτησε μια νομοθετική πρόταση ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, σαφήνεια και να μελετήσετε και να αξιολογήσετε αυτό το θέμα Τη διοσυνεργική διάσταση. Αυτή η πρόταση δεν αφορά τα μεγάλα φορτηγά οχήματα. Δεν έχουμε κάνει καμία μελέτη αντικτύπου για τη δημιουργία πανευρωπαϊκών προτύπων για μεγαλύτερα ε, οχήματα. Έχουμε, κα... έχουμε μελέτες, θετικές και αρνητικέ στα αποτελέσματά του αλλά έω τώρα. Εμείς ως Κομισιόν δεν έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία θέσπισης πανευρωπαϊκών προτύπων που να επιτρέπουν την κυκλοφορία μεγάλων, πολύ μεγάλων φορτηγών πανευρωπαϊκά. Και πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη έχουν αυτή την επιλογή στα χέρια τους. Το θέμα της Αυστρίας, που είναι η μάλλον πιο περίπλοκη χώρα εν προκειμένου, βλέπετε γεωγραφικά τη θέση της, ε, ότι είναι μια ορεινή χώρα, ε, φυσικά θα πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο ε, για την επικράτειά τη. Κατά πόσον επιτρέπει την κυκλοφορία τέτοιων μεγάλων οχημάτων ε, στους δρόμους της. Αν δεν θέλει, δεν θα κυκλοφορούν. <laughs> Okay. Just, um, you know, dear friends, it's, uh, you know... Αγαπητοί φίλοι, ε, ξέρετε, στην προηγούμενη θέση που είχα στην Κομισιόν μεταξύ άλλων κακών, ήμουν υπεύθυνο για, τα, για την κατασκευή κτηρίων και θυμάστε στον Περλεμόν μετά είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά. Τώρα άκουσα και αυτό το σήμα της πυρκαγιάς, που εντάξει είναι άσκηση, αλλά σε με αυτή την πυρκαγιά, μετά από αυτή την πυρκαγιά, άλλαξε η στάση όλων. Something is burning. No, no. And, and 2,000 people were... Uh, uh, Έγινε εκένωση 2.000 ατομών, αλλά αυτοεκένωση τόσο γρήγορα από το κτίριο που δεν είχα ξαναδεί τέτοια ταχύτητα. Λοιπόν, για τα giga liners, για τα πολύ μεγάλα φορτηγά οχήματα. Τα κράτη-μέλη έχουν αρκετή δύναμη να αποφασίσουν. Τρία κράτη-μέλη έχουν, επιτρέπουν, δύο κράτη-μέλη έχουν ξεκινήσει ε, δοκιμές και εγώ αν ε, βάλω το καπέλο του εκπροσώπου τοπικό, ε, τοπικής αρχής θα έλεγα ότι Και mm. uh, uh, Τεχνικά, αν το δείτε, αν λάβουμε υπόψη όλα τα τεχνικά στοιχεία, μπορείτε να μπείτε στο website της οργάνωσης των κατασκευαστών ε, οχημάτων, το ACA, και να δείτε και τη δική τους άποψη. Δεν είναι και αυτή τόσο σίγουροι ότι πάντοτε το βάρος συνδέεται αριθμητικά με το μέγεθος. κατασκευή των αξώνων, του σασί δηλαδή και των ε, ροδών. Δεν, δεν λειτουργεί πάντοτε έτσι. Και αυτή η πρόταση δεν έχει στόχο να επιτρέψει την κυκλοφορία, την πανευρωπαϊκή κυκλοφορία μεγαλύτερων φορτηγών. Είναι κάτι που εξέτασε νομικοί μας εμπειρογνώμονες. Ο νόμος, ότως ή άλλως, δεν το απαγορεύει αν ήδη δύο χώρε το επιτρέπουν, γίνεται η κυκλοφορία. Κάποιο ρώτησε έχει συγκεκριμένα. Ναι, ουσιαστικά μπορούν να διέλθουν ε, των σύνορων. Να μιλάμε για ένα σημείο